τον Ντάν Μαρή Κριστίν Βερζιά σχετικά με την εκστρατεία εμβολιασμού στι αναπτυσσόμενε χώρες. Υπάρχει πλέον για αυτή την γραπτή δήλωση η πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και επομένω, σύμφωνα και με το άρθρο 123 του κανονισμού ε, θα μεταδοθεί αρμοδίω και θα καταγραφεί στα πρακτικά. Πάρα πολύ σύντομα θα δώσω το λόγο στην κυρία Χόνεϊμπολ και στον κύριο Κέλλη για ελάχιστα δευτερόλεπτα στον καθέναν. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, γιατί υπογράψατε αυτήν την δήλωση. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ε, ε, πραγματικά είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που πέρασε το ψήφισμα αυτό, η δήλωση αυτή ε, που στηρίζει την εκστρατεία εμβολιασμού στις αναπτυσσόμενες χώρες με την Global Health Associates και με άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις εντός και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Είχαμε αγωνιστεί για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βερζιά, τον, την κυρία Ντεκεζέρ, τον κύριο Νιούτον Ντάρ και τον κύριο Κέλλη που θέλει να μιλήσει και εκείνο ο πρόεδρος. Ο κύριος Κέλλη. Κυρία Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα ε, θα ήθελα και εγώ να ε, ε, ευχαριστήσω όπως και η συνάδελφος Χόνιμπολ το κέρας της Αφρικής θα δεχθεί την γενεοδορία σας και αυτό σημαίνει δώρο ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Περνάμε τώρα στην έκθεση Καζάκ σχετικά με τις γενικές διατάξεις για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες. Τροπολογίες 1 ε, μέχρι 32, 34 μέχρι 53 on block υπέρ κατά